προβλέπεται εμείς σαν Επιτροπή να δουλέψουμε μέχρι τις 5. Μετά τις 5 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Μάρτιν, έχεις δει στο λόγο, όχι. Λοιπόν, σύντομη θα είναι η συνάντησή μας εδώ, γιατί στα πλαίσια των συντονιστών έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και ιδιαίτερα το θέμα της ε, πιθανής αλλαγής των συνθήκων. Ε, ε, λοιπόν, θεωρείται δεκτή η μερίσια διάταξη. Να σας μεταφέρω τις ανακοινώσεις. Ο συνάδελφος Μέσερ Σμιτ μας λέγει ότι η αρμόδια επιτροπή στο θέμα του είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και έχει αναβάλει την εξέταση της έκθεσης αυτής η έκθεση Wallis αναφέρομαι λέει ο Πρόεδρος και θα την συζητήσει τέλος Μαρτίου οπότε μπορούμε και εμείς να αναβάλουμε τη συζήτησή μας σύμφωνα με την πρόταση του κυρίου Μέσερ το Φεβράιο του 2012 26 Ιανουαρίου για την παρουσίαση των τροπολογιών. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα ήθελα να σα πληροφορήσω επίση ότι μετά από αίτημα της κυρίας Ρέγνερ και με τη συμφωνία του κυρίου Μέντες Δεβίγο ζητήθηκε να γίνει μια μελέτη από τη νομική υπηρεσία πάνω στα νομικά θέματα τα οποία τίθενται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βέβαια η γνωμοδότηση δεν έχει έρθει ακόμα, είναι στη φάση της επεξεργασίας και πρέπει να περιμένουμε. Ο συνάδελφος Γκαλτιέρη όπου να είναι φτάνει, έχει καθυστερήσει λίγο, και με παρακάλεσε αν είναι δυνατόν να αναβληθεί για αργότερα η συζήτηση του θέματος του, της εκθέσεως Νταφ μάλλον, της σχετικής με την ενιαία εκλογική διαδικασία. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τη συζήτηση εφόσον συμφωνεί και ο συνάδελφος Νταφ την έκθεσή του θα συζητήσουμε σε λίγο. Θα συζητήσουμε όμως πρώτα το επόμενο θέμα, το θέμα σε για τη μεταφορά σε πρωτόκολλο των δηλώσεων των σχετικών με την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δημοκρατία της Τσεχίας. Ο κύριος Μέντες Ντεβίγο που είναι υπεύθυνο για την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, ο Μέντες Ντεβίγο αλλά δεν είναι εδώ και πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε όμως εδώ τον κύριο Νταφ, όπως πάντα στην ώρα του ο κύριος Νταφ και γι' αυτό ε, θα μπορέσει να μας μιλήσει ο κύριος Νταφ αμέσως για το πρωτόκολλο ε, της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Δημοκρατία της Τσεχίας, τα θέματα 6 και 7 δηλαδή της ημερήσιας διάταξης ζητήθηκε γνωμοδότηση, η κυβέρνηση της Τσεχίας ζήτησε ε, το πρωτόκολλο μάλλον της Λισαβόνας, η συμπληρωματική συγγνώμη απόφαση για τη συνθήκη της Λισαβόνας να μετατροπεί σε πρωτόκολλο. Και αυτό πιθανώς μπορεί ε, το πρωτόκολλο αυτό να θεωρηθεί σαν... σε punti all'ordine del giorno che sono sostanzialmente collegati fra di loro. Σαν παράρτημα ή σαν συνημένο στην συνθήκη της Λισαβόνας. Ο κύριος Ντάφ, εν πάση περιπτώσει, έχει το λόγο να μας εξηγήσει. Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα σε όλους. Τα δύο σημεία που ζητείτε ως Ευρωκοινοβούλιο εμείς ε, να τοποθετηθούμε είναι πρώτον μια γνωμοδότηση επί της ουσίας όσον αφορά την δημοκρατία της Τσεχίας, την πρωτοβουλία της δημοκρατίας της Τσεχίας για την τροποποίηση των συνθήκων. Και δεύτερον από την άλλη πλευρά η λήψη απόφασης για το αν ή όχι θα συγκληθεί μια συντακτική συνέλευση και ίσως θα μπορούσα το δεύτερο σημείο να εξετάσω πρώτο. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να εμείνουμε και να επιμείνουμε στην σύγκληση μιας συντακτικής συνέλευσης. για να διαβουλευθεί επί της διαδικασίας αυτής. Και η δική μου άποψη επί της ουσίας όσον αφορά το αίτημα της Τσεχίας είναι μάλλον πιο επικριτική. Η τοποθέτησή μου πράγματι είναι ότι θα έπρεπε να ζητήσω ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην δεχτεί το αίτημα της πρότασης αυτής που υποβάλλει η Τσεχία και τα αναφέρω αυτά εν μέρη με τα θεμέλια ότι το πρωτόκολλο αριθμού 30 το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία μόνο τι ε, τίνος πρόκειται το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται νομική αβεβαιότητα και πολιτική σύγχυση τελικά μέσω μιας τέτοιας κατάστασης και τίποτα δεν θα μπορούσε να επανορθωθεί αν προσετίθετο και ένα τρίτο κράτος σε αυτά τα δύο, δηλαδή Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία που προανέφερα. Και πράγματι δηλαδή η επέκταση αυτών που δυνατόν, δυνάμει μπορεί να αποτελούν μια εν μέρη εξαίρεση από τη χάρτα αυτό θα ήταν, αν συνέβαινε, μια αποσταθεροποίηση, αποσταθεροποίηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη χρονική συγκυρία. και στο επεξηγηματικό υπόμνημα διερευνώ και εξετάζω τους λόγους για τους οποίους το σημερινό ενισχύ πρωτόκολλο θεωρώ ότι δεν βαίνει καλός και δημιουργεί προβλήματα. Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτοεξαίρεση από τη χάρτα εν τω μεταξύ αυτή η τοποθέτηση, αυτή η άποψη αμφισβητείται και από τους Βρετανούς νομομαθείς αλλά από την άλλη πλευρά και από το ίδιο το 10, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο. Και η πολωνική απόφαση πάλι να προσυπογραφεί αυτό το πρωτόκολλο ελήφθη για αντιφατικούς λόγους ελήφθη αυτή η απόφαση από τους Πολωνούς και τα πολωνικά δικαστήρια θεώρησαν καλύτερο να αγνοήσουν πλήρως αυτή τη συνιστόσα και μάλιστα πράγματι η Πολωνία, στην Πολωνία διεξάγεται ευρύτερη συζήτηση σήμερα για το αν θα έπρεπε ή όχι η Πολωνία να αποσυρθεί, να αποσύρει την υπογραφή της από το πρωτόκολλο αυτό. Από την άλλη πλευρά, στην Πράγα όπου βρισκόμουν την Παρασκευή σε σχέση με το επεξηγηματικό υπόμνημά μου για την περιγραφή ακριβώς της έκβασης ε, των συζητήσεων εκεί πώς είχε το πράγμα η ίδια η κυβέρνηση επιθυμεί να προχωρήσει γιατί θεωρεί ότι αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν τηρήσει τις υποσχέσεις του, αθετήσει τις υποσχέσεις του όσον αφορά την κυβέρνηση το Πολάνεκ, ε, τότε θα υπήρχε αντίδραση από πλευράς ε, του, των πολιτών, της κοινή γνώμης και κάποιοι εξέφρασαν επίσης τον φόβο ότι η δημοκρατία της Τσεχίας θα μπορούσε να αλλάζει τη γνώμη της και αποσυρώταν όσον αφορά την πρόταση αυτή, θα θεωρείται μια ανεύθυνη ή ένας μη αξιόπιστος εταίρος ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι αν υπήρχε ένα τέτοιο αίτημα για την απόσυρση αυτής της πρότασης από πλευράς της Τσεχίας, με μεγάλο σεβασμό θα αντιμετωπιζόταν και με ανακούφιση κιόλας. Είναι λοιπόν επίσης σαφές ε, όσον αφορά το Κοινοβούλιο της Τσεχίας ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται πλειοψηφία για την επικύρωση του πρωτοκόλου. Δεν είναι δεδομένη η αναγκαία αυτή η πλειοψηφία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κινούσαμε σε, με μια διαδικασία ε, διακυβερνητικής διάσκεψης ε, για την επικύρωση της, ε, του πρωτοκόλου. Και στο τέλος τέλος με την ανάληψη αυτής της ε, πρωτοβουλίας υπήρξε και άρνηση επικύρωσης. Θα μπορούσε να υπάρξει άρνηση επικύρωσης. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα όσον αφορά το δικαστήριο τις δικαστικές αρχές της Τσεχίας που σίγουρα είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ένα σενάριο στο οποίο θα υπάρξουν αιτήματα να τροχοπεδηθεί, να παγώσει το πρωτόκολλο. Τώρα, ο φόβος ή το αίτημα μάλλον το πρωτόκολλο όσον αφορά την Τσεχία ότι θα ρύθμιζε ή θα διασφάλιζε ότι τα διατάγματα μπένες δεν θα ξανά άνοιγαν ως θέμα νομίζω αυτό μπορεί να αρχιοθετηθεί και να θεωρηθεί πλέον ιστορικό γεγονός τσεχικός και ευρωπαϊκός και διεθνές, διεθνής νόμος, το, το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό και το τσεχικό δίκαιο τελεσίδικα καθόρισαν και σφράγισαν τα θέματα των διαταγμάτων Μπένες όταν η Τσεχία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι αυτά έχουν πλέον ρυθμιστεί και επειδή το Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι στεναρός υπέρμαχος της χάρτας και θα έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ως προπομπός, ως πρωτοπόρος για την προάσπιση της ακεραιότητας και της πλήρους εφαρμογής των αρχών αυτών πάντα σύμφωνα με την συνθήκη. Η δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να απορρίψουμε λοιπόν σαν συνέπεια όλων αυτών την πρόταση να ξανανοίξει το θέμα μιας διακυβερνητικής διάσκεψης ε, για αυτά τα θέματα. Φυσικά εμείς μόνο γνωμοδοτούμε, μια γνωμοδότηση υποβάλλουμε δεν είμαστε σε θέση να τροχοπεδίσουμε κάποια τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη. Όμως πρέπει να προσθέσω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα στην Πράγα με τα οποία είχα επαφές την Παρασκευή με κάθε τρόπο τόνισαν ότι το Ευρωκοινοβούλιο εδώ στις Βρυξέλλες θα έπρεπε να εκφράσει τις απόψεις του το ίδιο για αυτά τα θέματα τοποθετούμενο αναμφίσιμα, διότι υπάρχει ανάγκη να αποσαφινιστεί η θέση του Τσεχικού Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης για αυτά τα θέματα. Η Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου Πολιτικών Ελευθεριών, Επιτροπή ΛΥΜΕ, συντάσσει γνωμοδότηση γι' αυτό και θα έπρεπε να αναμείνουμε την υποβολή αυτής της γνωμοδότησης από πλευράς της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ προτού ψηφίσουμε. Όμως το χρονοδιάγραμμα που θα πρότεινα διαδικαστικά είναι να έχουμε υπόψη ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε κατά την συνεδρίασή μας του Ιανουαρίου και να περάσει το θέμα στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου. Δηλαδή όλα αυτά πριν από την κέρια σημασία συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο. σε σχέση με την απόφαση που θα ληφθεί να δοθεί συνέχεια ή όχι σε αυτό το ζήτημα και για να προσαφινιστούν αυτά απόλυτα θα δια... πρόκειται να διανύμω ένα επεξηγηματικό υπόμνημα στο άμεσο μέλλον τις επόμενες ε, δύο ημέρες ε, το αργότερο ώστε να δείτε πλήρως ε, πώς έχει η σύνοψη, η περίληψη αυτών των θέματων από πλευράς μου των συζητήσεων δηλαδή στην Πράγα Θεωρώ όμως ότι το υπόλοιπο του σχεδίου είναι ε, αυτοεπεξηγούμενο. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει διάφοροι το λόγο. Πάλα παρόλα. Α, ecco. <laughs> Prego, alla parola. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Νταφ που έχει τόσο σχολαστική προσέγγιση στο θέμα αυτό και μεγάλη πραγματογνωμοσύνη. Εγώ κατάγομαι από την Τσεχική Δημοκρατία και θα ήθελα μου επιτρέπετε να προσθέσω μερικές λεπτομέρειες οι οποίες προϋπήρχαν της όλης διαδικασία. Συμφωνώ, ομολογώ, ότι δεν θα πρέπει να συγκαλέσουμε συντακτική συνέλευση. Είναι πολύ μικρό το ζήτημα για να απασχολεί ολόκληρη συνέλευση, η οποία είναι για σπουδαία πράγματα προορισμένη. Επίσης συμφωνώ ότι θα πρέπει να απορρίψουμε το τσεχικό αίτημα. Να σας πω λοιπόν το ιστορικό. Όταν κυρώθηκε, μάλλον κατά τη δικασία της κύρωσης της ε, συνθήκης Λισαβόνας, ήμουν βουλευτής της Τσεχικής Βουλής και υπερψήφισα τη συνθήκη της Λισαβόνας χωρίς καμία πρόσθετη ε, προϋπόθεση ή όρο. Όπως και η Γερουσία κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα. Εκ των υστέρων μόνο ανέκυψε το αίτημα για ένα πρωτόκολλο χωρίς να έχει αυτό συζητηθεί σε κανένα σώμα του Κοινοβουλίου της ε, Τσεχικής Δημοκρατίας. Λοιπόν, τίθεται και το ερώτημα αν είναι συνταγματικό αυτό το αίτημα του πρωτοκόλλου κατά το τσεχικό σύνταγμα. Δεν θα το αναλύσω αυτό, ούτε αναλύθηκε επαρκώς. Και στη συνέχεια αποφάσισε η κυβέρνηση να καταθέσει το αίτημα για το πρωτόκολλο και η τσεχική γερουσία πλέον ενέκρινε ένα ψήφισμα που καλούσε την κυβέρνηση να αποσύρει το αίτημά της αυτό. Η τσεχική λοιπόν γερουσία ήταν υπέρ της απόσυρσης του αιτήματος για την αυτοεξαίρεση ή το opt-out. Δυστυχώς όμως η τσεχική κυβέρνηση συνέχισε σε αυτή τη γραμμή χωρίς ε, διαβούλευση με το Κοινοβούλιο Οπότε και δεν είναι γνωστή η θέση του Κοινοβουλίου. Συνοψίζω σύντομα ως εξή την κατάσταση. Πιστεύω προσωπικά ότι θα πρέπει να διακόψουμε τη διαδικασία, να την αναστείλουμε και να απευθυνθούμε στην Τσεχική Βουλή για να τη ρωτήσουμε πόσο πιθανή εκτιμάται την ε, κύρωση ενός τέτοιου αιτήματο. Θα ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια. Γιατί αν πέρασε από το Συμβούλιο και καταψηφιστεί στη Τσεχική Δημοκρατία, η κατάσταση θα είναι αρνητική. Μπραντς. Ευχαριστώ. Όταν υπέγραψε η συνήθιση της σαβόνας η Τσεχική Δημοκρατία, πίστεψα ότι υπέγραφε υπό τουλάχιστον ο πρόεδρος και ότι θα έχουν ε, μια διαφορετική σχέση με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, σε σχέση με, τα 24, με άλλα 24 κράτη δεν ε, χρησιμοποιώ το όρο opt-out, αυτό εξαίρεξη γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχο ε, τσεχικό ως όρος και αν χρησιμοποιήθηκε ποτέ και κυκλοφόρησε στον τύπο. Εάν θέλει η τσεχική δημοκρατία να συνεχίσει και να προωθήσει ακόμα αυτό το αίτημα, νομίζω ότι θα ήταν κακόπιστο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση να το απορρίψει. Δεν εναπόκειται σε εμά, στη τσεχική δημοκρατία, ε, να λέμε τι πρέπει να αποφασίσει, να αποφασίσουν εκείνοι. Και σε σχέση με το χάρτη, η Βρετανική κυβέρνηση το περιέγραψε αυτό ως αυτοεξαίρεση. Ξέρω ότι με διόρθωσε ο κύριος Νταφ και είπε Μπορεί η αγγλική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το ρόλο αυτοεξαίρεση opt-out, αλλά δεν είναι ουσιαστικά κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω δεν θέλω να σας ερμηνεύσω, αλλά θεωρείτε κύριε Νταφ ότι τα Βρετανικά δικαστήρια από ό,τι φαίνεται παρεμποδίζονται στο να ε, υλοποιήσουν αυτό το χάρτη σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα. Αλλά παραμένει ανοιχτό το ερώτημα. Κατά πόσο η Βρετανία ως κράτος θα μπορούσε να, να προσφύγει κάποιος εναντίον της στο δικαστήριο αν το πρωτογενές ε, δίκαιο έχει αμφισημίες. Ό,τι Ποια και να είναι η απάντηση όμως, νομίζω χρειαζόμαστε απάντηση. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου η σχέση δύο και ενδεχομένω ε, τριών ε, ε, κρατών με ένα σημαντικό έγγραφο όπω είναι η χάρτα αυτή είναι βέβαιη. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Δεν μπορούμε να αφήνουμε σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα να επικρατεί τέτοια αβεβαιότητα. Tak, Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Έχω δυσκολίες να καταλάβω καλά την νομική αξία και το νομικό βάρος που μπορεί να έχει το πρωτόκολλο το οποίο διαπραγματεύθηκε η Μεγάλη Βρετανία και η Πολωνία σχετικά με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να διευρύνουμε την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε άλλους τομείς, σε άλλα πεδία και στο πρωτόκολλο λέγεται ότι δεν υπάρχει άμεση υποχρεωτική εφαρμογή της χάρτας, οπότε δεν καταλαβαίνω την συμπληρωματική σημασία που αποδίδεται σε αυτό το πρωτόκολλο. Θα πρέπει παρόλα αυτά να σεβαστούμε το ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να θέτουν προϋποθέσεις για την επικύρωση εφόσον προχωρήσει η διαδικασία. Τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των εθνικών νομικών διαδικασιών αποφασίζουν για τις ε, συνθήκες με βάση τις οποίες αποδέχονται ή μη τη νέα συνθήκη. Νομίζω ότι αν εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίσουμε να ασχολούμεθα με πολιτικές συζητήσεις, οι οποίες βρίσκονται στη βάση των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, αυτό δεν θα ήταν καλό. Αν η κυβέρνηση της Τσεχίας ή μιας άλλης χώρας ε, επιθυμεί την ύπαρξη ενός τέτοιου πρωτοκόλου, δεν νομίζω ότι εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέμβουμε και να αποφασίσουμε για το υπέρ ή κατά της πρότασης. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Τσεχία, δεν ξέρω αν ο πρόεδρος, η Γερουσία, η Βουλή, η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν εμένουν στο αίτημα αυτό. Αλλά αν υπάρχει ένα κράτος μέλος το οποίο θέλει το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο θεωρεί σαν βάση για την σύνολη αποδοχή της συνθήκης, τότε σε αυτή την περίπτωση θα ήταν σοβαρό πολιτικό λάθος από πλευράς μας να αντιταχθούμε στο συγκεκριμένο αίτημα θα πρέπει να σεβόμεθα τις αποφάσεις των κρατών μελών, δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι και μπορούμε να ζητήσουμε από τις πολιτικές αρχές της Τσεχίας αν στο πρωτόκολλο και αν θα το δεχτούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Είναι θέμα καλών προθέσεων. Αν ε, θεωρεί κανείς ότι έχει υπογράψει ένα έγγραφο με βάση κάποια συνεννόηση και αυτή η συνεννόηση τροποποιείται, μπορεί να αποδυναμωθεί όλη εμπιστοσύνη στο σύστημα η Βρετανία θεώρησε ότι είχε υπογράψει την συνθήκη του Μάστριχτ με σαφείς ενδείξεις όσον αφορά και το χρόνο ε, εργασίας. Υπάρχει εδώ λοιπόν το θέμα του να τηρούν τον λόγο τους και τα υπεσχημένα τα κράτη-μέλη και ε, εδώ όχι με κάποιον περιορισμό Τώρα, για τη χάρτα, να υπενθυμίσω του συναδέλφου, του συναδέλφου, ότι υπάρχει και μια άλλη άποψη για αυτά τα θέματα. Κανεί δεν διαφωνεί με τις θεμελιώδεις αρχές της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θα βρείτε κανέναν Ευρωβουλευτή να διαφωνεί με την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συναθρίζεστε κτλ. Το πρόβλημα όμως είναι τα δημοκρατικά θέματα, αν κάποιο ε, λογοδοτεί έναντι ε, κάποιου ή όχι. Και θα δείτε παρόμοια θέματα σε σχέση με τα συντάγματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της πρώην Λαϊκή Δημοκρατίας της Ανατολικής Γερμανίας ε, και αυτά καθίστανται ανούσια και χωρίς περιεχόμενο όταν δεν υπάρχει δημοκρατικός μηχανισμός λογοδότησης. Τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα πρόβλημα με ε, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα με μαζικές ε, ε, εκτοπίσεις ή μαζικά φαινόμενα κατάσχεσης περιουσιών. Όμως οι πολίτες θεωρούν ότι έχουν αντληθεί οι εξουσίες από τους ερετούς εκπροσώπους που εκλέγουν οι πολίτες σε κάποιους γραφειοκράτες. Και αν συνεχίζουμε αυτή την πορεία μετάθεσης ευθυνών από τους πολιτικούς στους ανεύθυνους γραφειοκράτες, τότε δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μέντες Δεβίγο τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Νταφ για την εξαιρετική σου και λαμπρή παρουσίαση ε, του θέματος και του σχεδίου πρωτοκόλλου για το πώς θα εφαρμοστεί ο χάρτης αμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τσεχική Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εδώ ομιλούμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, ποια είναι η πραγματική αξία του πρωτοκόλλου παριθμών 30. Προς αυτή την κατεύθυνση ε, ήταν τα όσα είπε ο κύριος Δαφ. Είναι γεγονό ότι πολλές φορές οι πολιτικοί κάνουν κάποιες δηλώσεις έτσι κάπως απλουστευτικές των πραγμάτων και των καταστάσεων. Εγώ συμφωνώ από νομική απόψεω και ερμηνεία με τον κύριο Ντάφ ότι δεν είναι opt-out το πρωτόκολλο 30. Αλλά τι συμβαίνει, οι πολιτικοί για λόγου απλότητα και για να γίνουν κατανοητοί το ονομάζουν opt-out, αυτό εξαίρεση. Αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο. Επίση, θύμισε και ο κύριο Μέσσερ Σμιτ ότι αυτό δεν βρίσκει άμεση εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Αναφέρεται στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στι κυβερνήσει όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Είναι το άρθρο 51 του χάρτη που το είχε συντάξει ο κύριο Ρόμαν Χέρτσοκ, θυμάστε πρόεδρος τότε της συνέλευσης. Ε, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα λοιπόν. Και καλό είναι εδώ και συμφωνώ και με τον κύριο Μπρόνς να έχουμε και ένα ρόλο εμείς διαπαιδαγώγησης να εξηγούμε στους πολίτες τα πράγματα, να μην καταλαβαίνει κάθε πολίτης από το ίδιο κείμενο διαφορετικά πράγματα. Και έχω την αίσθηση ότι η έκθεση του κυρίου Νταφ προς αυτή την κατεύθυνση οδεύει. Εξηγεί ακριβώς ποια είναι η νομική αξία του πρωτοκόλου αυτού. Και νομίζω έτσι θα έχουμε συνεισφέρει πολύ ε, σε αυτή τη διαπαιδαγώγηση που με ενδιαφέρει και εμένα ιδιαίτερα. Και στο σημείο ΚΑΠΑ λατινικό ο κύριος Ντάφ εξηγεί πάρα πολύ καλά τι είναι το πρωτόκολλο 30. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα. Τώρα, κάτι τελείως διαφορετικό είναι αυτό που μας απασχολεί τώρα. Είναι η εφαρμογή, η διεύρυνση του πρωτοκόλλου αυτού προς την τσαχική δημοκρατία. Όλοι θυμούμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Ήταν η τελική απέτηση για να υπογράψει τη συνθήκη ο πρόεδρος της Οικικής Δημοκρατίας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορεί μένα να το βλέπουν κάπως και οι ιδέα αλλιώ, να το ονομάζουμε διαφορετικό τρόπο, αλλά περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πολιτικό ζήτημα που συνεδεύεται από πολλά παράδοξα. Όπως ε, ε, επισήμενε η συνάδελφος της Σοσιαλιστικής Ομάδας από την Τσεχική Δημοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λογικά βεβαίως, θα πρέπει να ε, σεβαστεί και να ανταποκριθεί στην υποχρέωση και που ε, ανέλαβε προς την Τσεχική Δημοκρατία. Και κάποια άλλη στιγμή, δεν ξέρω όταν ε, θα ενταχθεί η Κροατία, αλλά σε κάποια άλλη διαδικαστική στιγμή υποσχέθηκαν ότι θα ενσωματωθεί το αίτημα αυτό της τσεχικής κυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανταποκρίνεται στο καθήκον του. Όπως και για το Ιρλανδικό ζήτημα εντό εισαγωγικών που θα το δούμε στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Πάντα σύμφωνα με τη συνθήκη. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί αν συμφωνεί ή όχι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Νταφ, που μπορεί να σας φανεί ρητορική ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Κύριε Νταφ μου, τι θα συμβεί αν το Κοινοβούλιο αποφανθεί αρνητικά. Μπορεί να συνεχίσει, να δώσει συνέχεια στην πρόταση αυτή το Συμβούλιο. Γιατί μου φαίνεται ενδιαφέρον το θέμα. Ας πούμε ότι το Κοινοβούλιο πει εγώ δεν συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο θα μπορέσει, δικαιούται να προχωρήσει ή όχι. Ερωτώ τον κύριο Νταφ που είναι ειδικό εμπειρογνώμων και που ε, ήταν ήσυχο και ήρεμο ε, σήμερα το απόγευμα, του δώσω λίγη δουλειά ε, να δουλέψουν λίγο οι νευρώνε του και η φαιά του ουσία για να μην βαριέται. Λοιπόν, άλλο θέμα που παρά είναι επίσης παράδοξο. Το λέγουν όλοι, και ο κύριος Δαφ και οι σοσιαλίστρια συνάδελφος, ότι έχει έρθει η ώρα γιατί ε, χρειάζεται να ακυρώσουν και τα δύο σώματα του Τσεχικού Κοινοβουλίου και η Γερουσέλη ή όχι. Λοιπόν, και τι θα γίνει τώρα. Δεδομένου ότι είμαστε και σε περίοδο κρίσης και προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερες προσπάθειες και για να μην διονύζεται η διαδικασία, αν πούμε ότι ξέρουμε ότι δεν θα κυρωθεί και αν υπάρχει διαφορετική πλειοψηφία, τότε γιατί να μπούμε στη διαδικασία αυτή από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες πώς έχουμε εμπλακεί σε αυτή την ιστορία με τις κυρώσεις, τις επικυρώσεις, τα κοινοβούλια και με τα ίδια η κυβέρνηση που το ζήτησε δεν συμφωνεί ε, με το κοινοβούλιο της και καταψηφίζει τι είναι αυτά τα πράγματα περίεργα. Και ένα τελευταίο. το λεγόμενο δικαίωμα ε, του βέτο ή της ε, ανησυχηρίας και την ομοφωνία. Ιδού ένα καλό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί με τρόπο διεστραμμένο αυτή η ιστορία. Διότι εκείνοι που υποστηρίζουν το βέτο λένε ότι ορίστε θα έχω το δικαίωμα να βάλω βέτα μου δεν μου αρέσει κάτι. Ναι. Αυτό όμως το δικαίωμα το έχουν και οι υπόλοιποι 26, όχι μόνο εσύ και οποιοδήποτε άλλο εθνικό κοινοβούλιο θα μπορούσε να μην επικυρώσει αυτό το πρωτόκολλο. Και έρχομαι στην επόμενη μου σκέψη, κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα είπαμε, λέμε και πάλι ότι θα υπάρξει αναθεώρηση της συνθήκης, τουλάχιστον το συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία αναφέρεται αυτό της Τσεντεού και τα γράφει σήμερα ο τύπος. Αν γίνει αυτό, χωρίς δημογωγία καμία, με κοινή λογική, Ε, παραλίγο να πω όπως αρμόζει, όπως θέλει ο Θεός, αλλά με αγριοκοιτάει ο κύριος Γκερέρο. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε με κανονικό τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ε, μια εναλλακτική φόρμουλα ε, για να παρακάμψουμε κάπως την ομοφωνία, γιατί η ομοφωνία είναι διπλής κατεύθυνσης. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι ε, εγγύηση για να μην επιβάλλει κανένας τίποτα σε κανέναν άλλο. Αλλά μπορεί οποιοδήποτε άλλος να βάλει βέτο σε μια Ευρώπη των 27 όπου ζητούμε προστιθέμενη αξία, ταχύτητα δράσης, αποτελεσματικότητα, έχω την αίσθηση ότι είναι μέγας αναχρονισμός η ομοφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μέντες Δεβίγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γουερέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. όλοι οι παρόντες διαπίστωσαν ε, την ε, εξωφρενική ευγλωτία και τον ενθουσιασμό του κυρίου Μέντες Δεβίγο που οφείλεται σε ένα ανθρωπολογικό ενθουσιασμό που αν δεν γνωρίζετε τα πράγματα απορρέει από την εκλογική τους νίκη στην Ισπανία. Συγχαρητήρια προσωπικά και σε εσά και στο κόμμα σας και έχει αφήσει τώρα στενό περιθώριο, σαν αυτό που πήραμε χτες οι Ισπανοί οι για να πω και εγώ δύο λόγια. Θα ήθελα όμως να τονίσω τα εξή τρία θέματα, τα οποία εξέτασε και ο ίδιος. Το πρώτο έχει να κάνει με ε, την αφετηρία και την αφορμή του θέματος αυτό, το δεύτερο εσωτερική κατάσταση ε, στην Τσεχία και ε, ε, το τρίτο θέμα είναι πώς συνδέεται με τρόπο έτσι στρεβλωμένο με την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο λοιπόν, ποια είναι η προέλευση και το ιστορικό, το γνωρίζουμε. Ένας πρόεδρος ενός κράτους μέλους της Ένωσης ενώ το κοινοβούλιο του ήταν υπέρ, εκείνος μέχρι τη τελευταία στιγμή φρέναρε την υπόθεση αυτή και την κύρωση της ένδειξης Λισαβόνας και έκανε μία εμφάνιση ε, όχι μόνο με δηλώσεις αλλά και με κάποια έπαρση έτσι ότι εγώ θα υπογράψω αλλά τι θα μου δώσετε για να υπογράψω. Και αυτό δείχνει ότι είναι βαθιά αντιευρωπαϊστής. Γιατί το να κάνει κανείς τέτοιες δηλώσεις για υποτιθέμενα ή πραγματικά δικαιώματα κάποιου πληθυσμού ή κάποιου λαού σε κάποια άλλη ιστορική στιγμή της ε, Ένωσης, ε, της οικοδόμησης, που ανήκει όμως στο παρελθόν, το ιστορικό. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την εσωτερική κατάσταση και το ίδιο το κοινοβούλιο της Τσεχίας γιατί έχει διαφορετική πλειοψηφία το κάθε σώμα αλλά πρέπει να κυρωθεί και από τα δύο σώματα η συνθήκη και υπάρχει το ενδεχόμενο να μπούμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία που είναι αρκετά δεδαλώδης και μετά μπορεί να έχουμε την εξής κατάσταση το είπαν και πολλοί προαρίσανες εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε και μια εσωτερική συνεδρία συγκλειστή και μας ε, το ανέφερε ένας εκπρόσωπος της πλειοψηφίας στη Γερουσία ότι μπορεί να οδηγηθεί σε εμπλοκή εσωτερικά αυτή η διαδικασία. Ενώ εμείς θα έχουμε ξεκινήσει κατόπιν αιτήματος της ίδιας της χώρες που τώρα το μπλοκάρει. Και το τρίτο θέμα από πολιτικής απόψεως ενδεχομένως να είναι πιο περίπλοκο, αλλά και, πώς να το πω, πιο καταστροφικό ταυτόχρονα. Ότι αυτό το θέμα μπορεί να δυσκολεύσει, να εμποδίσει, να οδηγήσει σε ομοιρία την ένταξη της Κροατίας. Μπορεί να φαίνεται ότι έχει αρχίσει η διαδικασία για να διαχωριστούν αυτά τα δύο, Έχω την αίσθηση ότι μία από τις ανησυχίες που αναφέρει στην έκθεσή του ο κύριος Νταφ είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια στεναρή στάση εδώ λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να συνδέουμε την επίλυση του θέματος αυτού με την ένταξη της Κροατίας και Τούμπαλιν. Είναι δύο ανεξάρτητα θέματα γιατί αυτό το θέμα ας πούμε, μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα, αλλά να προχωρήσει το θέμα της Κροατίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κύριε Γκουερέρο. Δεν υπάρχουν άλλοι βουλευτέ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Νταφ θέλει να αντιδράσει στις προτάσεις που ακούστηκαν. Μπορεί να το κάνει τώρα. Είμαι ε, ε, λοιπόν σε όσους πήρε το λόγο, στον κύριο Μπρόντς. Θα ήθελα να πω ότι η Βρετανική θέση κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια μορφή ακρεμότητας. Το εφετείο ήρθε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και ζήτησε μια γνωμοδότηση για την έννοια, για το νόημα μάλλον, του πρωτοκόλου. Πρόκειται για τη λεγόμενη περίπτωση ΣΑΙΝΤΗ από το όνομα κάποιου που ζήτησε πολιτικό άσυλο και ο οποίος παραπονείται ότι παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Δεν μιλάμε για μαζική για μαζικό εκτοπισμό πληθυσμών, αλλά για μία συγκεκριμένη περίπτωση. Η βασική αρχή η οποία εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να απορρίψει ουσιαστικά την ισχύ του πρωτοκόλου σε σχέση τουλάχιστον με τη συγκεκριμένη περίπτωση ΣΑΙΔΗ και λέγει ότι τα Βρετανικά δικαστήρια ήταν απολύτως ελεύθερα να δεχθούν τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος σε σχέση με την ισχύ ε, του, ε, ε, της χάρτας. Η τελική κατάληξη για την απόφαση του δικαστηρίου ε, δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι, αλλά παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι πάνω κάτω το δικαστήριο θα ακολουθήσει την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα. και οι απόψεις των αρμοδίων και η νομολογία και στην Μεγάλη Βρετανία και στην Πολωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούν. Νομίζω ότι έχουμε πλέον αρκετή εμπειρία από την εφαρμογή της, κάρτα, της χάρτας συγγνώμη, σαν δεσμευτικό νομικό κείμενο, σαν νομικό μέσο πλέον και έτσι μπορούμε εμείς πολιτικά να πούμε κάλλιστα ότι το πρωτόκολλο αυτό είναι κάτι το θετικό ή, ή αντίθετα αν δεν συμφωνούμε είναι κάτι το αρνητικό. Νομίζω ότι καθήκον μας πλέον είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία μορφή προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη οι εξαιρέσει, οι αποκλήσεις οι οποίες στοχεύονται στη συγκεκριμένη περίπτωση από το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και στηρίζονται από αυτό δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση τον σεβασμό αυτό. Τώρα δεν ξέρω εγώ, δεν θα πω εγώ τι θα πρέπει να κάνει η Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά έχει σημασία να καταλήξουμε σε μια αυτόνομη αντίληψη αντίληψη η οποία να μην εκφράζει μόνο την προοπτική την οποία έχουν στο συγκεκριμένο θέμα οι Τσέχοι αλλά και συνολικά τις απόψεις τις οποίες έχουν όλα τα κράτη-μέλη και οι λαοί που τους συναποτελούν. Ο Μέντες Δεβίγος νομίζω ότι απέκλεινε κατά τη διάρκεια της εξαιρετική πρότασης την οποία έκανε από τη συνθήκη και ζήτησε να καταστεί το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης πρότασης ευρύτερο. Σε αυτό δεν διαφωνώ. αν μου ζητήσετε να σας πω ποια θα είναι η απόφαση, η αντίδραση του Συμβουλίου στην περίπτωση κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει με την γνωμοδότησή του την πρόταση, τότε πράγματι η απάντηση θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορώ να την πω. Νομίζω ότι το Συμβούλιο θα καθοδηγηθεί από τις ε, απόψεις του Τσέχου Πρωθυπουργού uh, και η τσεχική κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει αν θα εμείνει ή όχι. για να καταλήξει στην τελική απόφαση θα πρέπει να προσμετρήσει την περιπλοκότητα των τσεχικών κοινοβουλευτικών απόψεων και των απόψεων των ανωτάτων συνταγματικών δικαστηρίων της χώρας. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Συνεπώς, εφόσον θέλουμε εμείς να ψηφίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου, η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών θα είναι η Δευτέρα Φεβρουαρίου. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό ε, νωρίτερα, τότε στις 25. Κοιτάξτε, λέει ο κύριος Νταφ. Εγώ κάνω την πρόταση να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο σε επίπεδο επίτροπή στο τέλος του μηνός Ιανουαρίου. Ναι, αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση, αυτήν θα σας παρουσίαζα. Προβλέπει λοιπόν ψηφοφορία στις 25 Ιανουαρίου με προθεσμία κατάθεση τροπολογιών την 15η Δεκεμβρίου. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρείται ότι συμφωνήθηκε. Λοιπόν, έχουμε και το Μέντερ Δεβίγου ανάμεσά μας passo indietro e illustrarci il tema del protocollo και μπορεί να μας παρουσιάσει τις ανησυχίες του για το πρωτόκολλο το σχετικό με τις Ιρλανδικές θέσεις γύρω από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και εδώ έχουμε δύο εκθέσεις μεθοδολογικά διαφορετικού περιεχομένου και τις δύο θα τις αντιμετωπίσει ο κύριος Μέντες από κοινού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι το απόγευμα των πρωτοκόλων. Αλλά είναι διαφορετική η φύη των δύο πρωτοκόλων. Ο κύριος Γκερέιρο είπε πολύ εύγλωτα ότι η διεύρυνση του πρωτοκόλου περιθμών 30 προς την Τσεχική Δημοκρατία ήταν απέτηση τελευταίας στιγμής στο παραπέντε για να υπογράψει ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα παραπάνω στα όσα είπε ο κ. Δέρα. Τώρα έχουμε όμως μια διαφορετική περίπτωση. Θα προσπαθήσω να σας εξιστορήσω σε συντομία το τι συνέβη. Όπως γνωρίζετε, η Ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει σε δημοψήφισμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Εγώ θυμάμαι εκείνη την εποχή πόσο επίμαχο ήταν το θέμα στο Κοινοβούλιο για το κατά πόσο ήταν υποχρεωτικό ή όχι αυτό το δημοψήφισμα. Θυμάμαι ο κύριος Ντάφ και εγώ είχαμε ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση για το εάν όντως η Ιρλανδική κυβέρνηση ήταν ε, από τον νόμο υποχρεωμένη να κάνει δημοψήφισμα ή όχι. Και λέγαμε ότι όχι, αλλά εν περιπτώσει το έπραξε δικαίωμά τη και το έκανε. Στο δημοψήφισμα λοιπόν αυτό, όπου μερικοί συμμετείχαμε, ίσως δεν θα έπρεπε να το πω γιατί ήταν ε, το αποτέλεσμα αυτό που ήταν, μερικοί περασπιστήκαμε το ναι, βγήκε το όχι. Λοιπόν, όπως συμβαίνει πάντα, η κυβέρνηση που υπέβαλε σε δημοψήφισμα μια συνθήκη της Ένωσης, που είχε ήδη διαπραγματευτεί και υπογράψει δεν μπορούσε να κυρώσει. Οπότε αυτή η κυβέρνηση ψάχνει μια διέξοδο συνήθω. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές αυτό που μένει, αυτό που ορισμένοι ε, διηγούνται είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στη χώρα αυτή να κάνει και δεύτερο δημοψήφισμα. Εγώ δεν κατηγορώ καθόλου την κυβέρνηση της Ιρλανδίας, αλλά ήρθε ο Πρωθυπουργός ο φίλος Μπέρτι Αχιάρν, αν θυμάμαι καλά τότε. Λοιπόν, το είπαμε. Λοιπόν, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, εσύ θέλησε να το βάλεις σε δημοψήφισμα. Βγήκε το όχι. Τώρα τι θα κάνεις, αγαπητέ μου. Δεν, δεν του λέμε κάνε δεύτερο δημοψήφισμα. Του λέμε πώς θα βγεις από αυτό το αδιέξοδο τώρα. Ο κύριος Αχιάρν κάτσε, το σκέφτηκε και μετά από λίγο καιρό νομίζω μεσολάβησαν και εκλογές και βγήκε άλλος πρωθυπουργό, ο κύριος Κόουεν, αποφάσισαν, εν πάση περιπτώσει, οι Ιρλανδοί, αφού ανέλησαν τους λόγους γιατί οι Ιρλανδοί καταψήφισαν τη συνθήκη, αποφάσισαν τα εξή δύο. Πρώτον, κάτι που δεν είναι στην έκθεσή μου και δεν θα αποφαθούμε γι' αυτό, να απαλληφθεί η διάταξη τη συνθήκη τη Λισαβόνα που ήρθε από τη διακυβερνητική γύρι στο επαρόδο διάσκεψη και όχι από την κοινοβουλευτική συνέλευση που έλεγε να είναι λιγότερη επιτροπή από τον αριθμό των κρατών και ορισμένοι από εμάς πραγματικά λυπούμεθα για αυτή την κατάσταση ότι θα πρέπει οπωσδήποτε κάθε χώρα να έχει τον επίτροπό της. Αυτό νομίζω ότι είναι βαθιά λανθασμένο ως αντίληψη. Εν πάση περιπτώσει θεώρησαν οι Ιρλανδοί ότι και ήταν ένα από τα επιχειρήματα, το θυμάμαι πολύ καλά, της εκστρατείας του όχι, θεώρησαν ότι ήταν προαπαιτούμενο να υπάρχει πάντα Ιρλανδός Επίτροπος. για να κατανοούν οι Ιρλανδοί ότι είναι θετική συνθήκη. Αυτό όμως δεν είναι το παρόντος. Ήταν μια πολιτική συμφωνία εγώ κάνω μια πολιτική αξιολόγηση ότι δυστυχώς έχουμε ένα επίτροπο αναχώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκτός αυτού όμως, και επιμένω, αυτό δεν μας ε, απασχολεί, δεν μας ζητούν αυτό. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ζήτησε διευκρίνηση, λέει, ερμηνεία διευκρινιστική ορισμένων διατάξεων της συνθήκης της Λισαβόνας που είχαν προκαλέσει μια αντιπαράθεση στη συζήτηση πριν το δημοψήφισμα. Τι εννοώ. Οι πολέμοι της συνθήκης είχαν πει ότι η συνθήκη λέει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν λέει. Λοιπόν, τι ζητάει η Ιρλανδική κυβέρνηση από το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ερμηνεύστε αυτά που λέει η συνθήκη για να μην παρερμηνεύετε από τους πολέμιους του δημοψηφίσματος. Ελπίζω να το είπα καλά το γλωσσοδέτη, γιατί γλωσσοδέτης είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το δέχθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει τι ορίζει η συνθήκη και να την ερμηνεύσει. Η Ιρλανδική κυβέρνηση εξέτασε, μελέτησε αυτές τις δυσκολίες στην Ερμηνεία, για να το πω ε, εύσχημα, και ε, τις έχει χωρίσει σε τρεις μεγάλες ενότητες. Το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια και την παιδεία, το ένα κεφάλαιο. Το δεύτερο είναι η φορολογία και το τρίτο είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Το πρωτόκολλο που ενέκρινε λοιπόν το Συμβούλιο ως απόρρια εκείνης της απόφασης που είχε λάβει το μήνα Ιούνιο αν δεν απατώμε του 2009 ήταν επεξημαγητική και εξήγησε ότι καμία διάταξη δεν πρόνοια της συνθήκης που έχει σχέση με το χάρτη λιδών δικαιωμάτων δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι θίγει το δικαίωμα στη ζωή όπως ορίζεται από το Ελλαδικό Σύνταγμα ή τα δικαιώματα στη, για την οικογένεια, για την παιδεία, για την εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι θέματα του Ελλαδικού Συντάγματος. Βεβαίως ισχύει αυτό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ομοθετεί για τα δικαιώματα στη ζωή και για την παιδεία έχει μόνο συμπληρωματική ε, αρμοδιότητα. Ξεκαθαρίστηκε λοιπόν αυτό. Άλλο θέμα τώρα φορολογία. Θα ήθελα εδώ να ακούσω τις απόψεις σας, διότι έχω την αίσθηση ότι το σχέδιο πρωτοκόλλου στη διατύπωσή του είναι κάπως απόλυτο. Δεν υπάρχει πουθενά στη συνθήκη της Λισαβόνας καμία αλλαγή ε, για κανένα κράτος μέλος σε ό,τι αφορά τα φορολογικά θέματα. Αυτό είναι έτσι βαριά δήλωση, πάρα πολύ ισχυρή. Δεν είμαι βεβαίως ότι ισχύει αυτό ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σας αναφέρω και τις δικές μου ανησυχίες. Και για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, είναι το πιο μακροσκελές άρθρο, δεν σας το διαβάσω, το έχετε. Αλλά σε αυτά τα θέματα της ασφάλειας και άμυνας, πρώτον, δεν θίγεται η παραδοσιακή ουδετερότητα της Ιρλανδίας και δεύτερον, όλα αυτά τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και ενδεχομένω να την αφορούν, θα πρέπει να ληφθούν ε, τη συμφωνία της ε, Ιρλανδίας. Αν δεν συμφωνεί η Ιρλανδική κυβέρνηση, δεν λαμβάνονται τα μέτρα αυτά. Αυτό έχει να κάνει με τη διαρθρωμένη συνεργασία. Λοιπόν, με την επιφύλαξη που αναφέρω για τη φορολογία, γιατί νομίζω ότι τα λέει πολύ απόλυτα και δεν ισχύουν έτσι. Όλα τα υπόλοιπα, τι είναι. Έρχεται το πρωτόκολλο και εξηγεί τι λέει η συνθήκη. Και τίποτα παραπάνω. Συνέπεια αυτή τη δήλωση ήταν η δυνατότητα που δόθηκε στην Ιρλανδική κυβέρνηση να προχωρήσει. Αφού είχε εξασφαλίσει τον Επίτροπο και αφού είχε διευκρινίσει αυτά τα θέματα, έκανε και δεύτερο δημοψήφισμα το οποίο δέχθη τις ευλογίες του Ιρλανδικού λαού και προχώρησε η κύρωση και η σε ισχύ της συνθήκης. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τώρα έχει έρθει η ώρα να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα η Ιρλανδική κυβέρνηση έκανε εκείνο που της αναλογεί και το συγκεκριμένο πρωτόκολλο δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να εξηγεί τι λέει η συνθήκη. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα κύριε Πρόεδρε να προχωρήσουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να συγκαλέσουμε συνέλευση για να εγκρίνουμε αυτό το πρωτόκολλο. Μπορούμε να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας και το μόνο που κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε στα όσα συμφωνήσαμε σε εκείνη την ε, προϋπόθεση και το προαπαιτούμενο για να γίνει το δεύτερο δημοψήφισμα. Σε αντίθεση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, για τους λόγους που εξήγησε ο κύριος Νταφ, νομίζω ότι εδώ δεν έχει τίποτα που να επηρεάζει τα δικαιώματα των Ιρλανδών ούτε κανενός άλλου Ευρωπαίου πολίτη. Ε, άρα λοιπόν, όχι στη σύγκληση τη διδακτικής συνέλευση, και ναι ε, στη σύμφωνη γνώμη υπέρ του πρωτοκόλλου. Ευχαριστώ. Okay. Είχε ζητήσει πρώτο το λόγο ο κύριος Μάρτιν και μετά ο κύριος Νταφ. Νομίζω ότι τα πρωτόκολλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια χρόνια ουσιαστικά μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης και μας κάνουν να σκεφτούμε το πώς εφαρμόζονται οι προβλέψεις της συνθήκης. Θέλω να επιστρέψω τα συγχαρητήρια τα οποία Απίθυνε προς εμέ ο κύριος Δεβίγο. Η συνέπεια αυτής της συμφωνίας ήταν ένας επίτροπος ανακράτος, το οποίο μπορεί κάποια φάση να αλλάξει, αλλά όχι όμως σε αυτή τη φάση. Συμφωνώ με τον εισηγητή απόλυτα ότι το άρθρο 2 Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή όπου υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνει συντακτική συνέλευση και διακυβερνητική είναι κάτι το οποίο θα αυξήσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φορολογίας. Το άρθρο 2 του Ιρλανδικού πρωτοκόλου ε, φαίνεται λίγο περίεργο στη συγκεκριμένη φάση. και νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα επιβιώσει επί μακρόν. Σχετικά με το άρθρο τώρα, μιας και δεν φαίνεται ότι θα ξεσπάσει πόλεμος όπου να είναι, είναι κάτι το οποίο δεν θα δημιουργήσει καμιά ιδιαίτερη διαφορά ούτε για τους Ιρλανδούς ούτε για μας. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι συλλαμβάνω αυτό το οποίο θέλει ο εισηγητής. Από την άλλη δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε κριτική στα πλαίσια των αιτιολογικών σχέσεων της ποιότητας του πρωτοκόλου αυτού και των διαδικασιών που οδήγησαν σε αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα πλέον ήρθε η σειρά του κυρίου Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ομιλώ εκ μέρους του κυρίου Μορέιρα, ο οποίος είναι ο σοσιαλιστής, ε, ο σκιώδης μάλλον εισηγητής μας. Μου έστειλε ένα μικρό σημείωμα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία έχω από τον κύριο Νταφ, άκουσα από τον κύριο Νταφ και τον κύριο Μέντες Δεβίγο. Μπορεί να πει κανείς ότι το πρωτόκολλο αυτό απέκτησε δεσμευτικά νομικό καθεστώς άμα τη θέσει σε ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνα. Οπότε είναι πάρα πολύ περίεργη η συζήτηση την οποία κάνουμε σε αυτή τη φάση. Ο καθηγητής συμφωνεί λοιπόν με τον εισηγητή ότι η πρόταση για το πρωτόκολλο είναι πλήρως συμβατή με τις συνθήκες και στην ουσία καθιστά περισσότερο κατανοητό το περιεχόμενο της συνθήκης. Πρόκειται για μια δήλωση η οποία διασφαλίζει τους Ιρλανδούς πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία που οδήγησε στο δημοψήφισμα. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας και γι' αυτό δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήματα για μας. Και ο καθηγητής Μωρέιβε δεν έχει καμία διαφωνία να προχωρήσουμε ε, μέσα από το πρωτόκολλο και στην ένταξη της Κροατίας. Κύριος Μπρόντς. Κύριος Μπρόντς. Σχετικά με τις ανησυχίες των Ιρλανδών γύρω από τη συνθήκη Αυτές θα έλεγα έχουν σαν στόχο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όχι το Συμβούλιο γενικότερα και δεν ακολουθήθηκαν οι αποφάσεις αυτές από νομοθετικές ρυθμίσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι νομοθετικό σώμα και σχετικά τώρα με αυτά τα οποία υποστήριξε και η τσεχική δημοκρατία και αυτά δεν προκάλεσαν επιπλέον νομοθετική παραγωγή θα έλεγα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το θέμα είναι ότι και στην περίπτωση της Ιρλανδική, την Ιρλανδική και στην περίπτωση της Τσεχίας η πρόταση αυτή έχει γίνει αντικείμενο επικύρωσης από 26 ε, χώρες. Συγγνώμη αν εκθέτω εδώ κάποιους, αλλά εφόσον έχουν ήδη ε, γίνει αντικείμενο υπογραφής και επικύρωσης, τότε τι νόημα έχει το πρωτόκολλο αυτό με τέτοια καθυστέρηση. Διερωτώ με αν είναι ή ήταν το πρωτόκολλο νομικά δεσμευτικό. Προφανώς όχι. Κύριε Μέντε Δεβίγο, μπορείτε να δώσετε απαντήσεις. Μια πολύ σκόπιμη συζήτηση και ευχαριστώ να απαντήσω. Και προηγούμενα ευχαριστώ τον κύριο Ντάφ για την παρέμβασή του και πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα ότι στα σκεπτικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, κυρίως μια αναφορά στο θέμα δηλαδή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε. Είναι ένα θα ήταν ένα μεγάλο πολιτικό σφάλμα. Ωστόσο όμως είναι ένα θέμα το οποίο δεν ε, εντάσσεται στο θέμα του πρωτοκόλλου. Και πάλι το τρίτο, ασφάλεια και άμυνα. Θα το εξετάσω και αυτό με πολύ προσοχή με μια πρώτη ανάγνωση που έκανα μου φαίνεται ότι συνάδει με τη συνθήκη αλλά θα το ξαναδώ με ιδιαίτερη προσοχή και όσον αφορά τη σοσιαλιστική ομάδα τον ε, κύριο Μάρτιν, τον ε, καθηγητή ε, Βιτάλ Μορέιρα, συμπίπτω με την άποψή τους ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να επιλύσουμε ένα πολιτικό θέμα, μια πολιτική απόφαση από πλευρά του Συμβουλίου και όχι νομοθετική. Και αυτό είναι η πολιτική επίπτωση και γι' αυτό πρέπει σε σχέση με το πρωτόκολλο που έχει ταυτόσιμη ε, σημασία με, το, με τη συνθήκη θα πρέπει να υποβληθεί προς επικύρωση στα 27 κοινοβούλια. Θεώρησε η κυβέρνηση της ε, Ιρλανδίας ότι η πολιτική απόφαση επαρκούσε σε σχέση με την ε, ερμηνεία αυτή της συνθήκης και προσφυγή σε ένα δημοψήφισμα. Αυτό που κάνουμε κατά κάποιο τρόπο είναι να τηρήσουμε τα συμπεφωνημένα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και πάλι επιμένω εκτός αν υπάρχουν κάποιες ε, εξαιρέσεις ή εξαιρετικές περιπτώσεις όπως της Τσεχίας, θα πρέπει τα υπεσχημένα να τηρούνται. Και θα δίνουμε μια νομική ε, εξουσία στο πρωτόκολλο που νομίζω ότι δεν έχει αφέ αυτού. Ε, Καλώς μου φαίνεται λοιπόν ότι μπορούμε να ορίσουμε την 25η Ιανουαρίου για την παρουσίαση και την ψηφοφορία στις 28 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως, σημειώνοντας ότι πράγματι η δήλωση σχετική για την Ιρλανδία έχει μια ερμηνευτική ιδιότητα και πόσο μάλλον το άρθρο 2 ακριβώς αυτό διευκρινίζει. Και λέγεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει τίποτα στη συνθήκη για οποιοδήποτε κράτο μέλος και όχι μόνο για την Ιρλανδία. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 3, το σχετικό με την ασφάλεια και άμυνα. Δεν τροποποιείται τίποτα, απλά ενισχύεται το αντίστοιχο άρθρο της συνθήκης. Και η έκφαση για οδήποτε κράτος μέλος δεν αφορά περιπτώσεις όπως τον Ευρωπαϊκό Κοινό Στρατό, σαν παράδειγμα, αλλά είναι αυτονόητο είναι ότι είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν προκαταλαμβάνει αυτό που ορισμένοι θα ήθελαν να ονομάσουν ε, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Έχει μία θα έλεγα σημασία αυστηρά ερμηνευτική. Η συζήτηση θα γίνει όμως μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, όπου θα παρουσιαστεί επίσημα και θα ψηφίσουμε 28 Φεβρουαρίου. Θα πάμε ακόμα πιο πίσω ανάποδα σήμερα και θα αντιμετωπίσουμε την έκθεση DAF για την ενιαία εκλογική διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν γίνει συζητήσεις, έχει απορριφθεί το πρώτο σχέδιο, έχει παρουσιάσει ένα δεύτερο σχέδιο από τον εισηγητή Έγινε μια πρώτη συζήτηση μέχρι τις 27 Οκτωβρίου κατατέθηκαν τροπολογίες από Βίλαν Σέφλιν, Κόξ, Λαμασούρ, Σόντεργαρντο, Σούλτς, Χάκλαντ και άλλους. Μπορούμε να συζητήσουμε από σήμερα αν θέλετε αυτές τις τροπολογίες. Θα έλεγα ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη έκθεση και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλά τι διαδικασία θα ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξή. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει ζητήσει το λόγο αργότερα να πάρει το λόγο ο κύριος Γουαλτιέρη αλλά δεν μπορούμε άλλο να καθυστερήσουμε και δίνουμε το λόγο στον κύριο Νταφ. Μάλιστα. Όπως είπατε, 40-45 τροπολογίες είχαμε που εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες ουσιαστικά. Η πρώτη ήταν εκείνες που καταρχήν απορρίπτουν την ιδέα μιας πανευρωπαϊκής ε, τέτοιας προσέγγισης ε, και πολυεθνικών τέτοιων πινάκων και θα είμαι κατά στην ψηφοφορία αυτών. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνες που δεν είναι απόλυτα σαφείς και κάνω λόγο εδώ για τις τροπολογίες του κυρίου Βίλαντ και του κυρίου Σούλτς ιδιαίτερα που έχουν καλές προθέσεις χωρίς καμιά αμφιβολία σίγουρα όμως δεν επαναλαμβάνω, δεν βελτιώνουν την σαφήνεια του ψηφίσματος, του κειμένου του ψηφίσματος. Και μια τρίτη κατηγορία τροπολογιών και εδώ ο Ρομπέρτο Γκουαντιέρη μόλις έφτασε, βλέπω, καλό σας απόγευμα. Βρίσκω ότι Κάποιες από αυτές θα μπορούσα να τις ε, δεχτώ με κάποια μικρή τροποποίηση στη διατύπωση, όμως ωστόσο δεν θα ήθελα να περιπλέξουμε τα πράγματα υπερβολικά. Για παράδειγμα, σε σχέση με την δεύτερη έκθεση, το νόημα ήταν στην παράγραφο 11 να υπάρξει μία ατζέντα για τον διάλογο με το Συμβούλιο. τα πράγματα με τα οποία δεν μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο να συμφωνήσει άμεσα επ' αυτών. Και θα προτιμούσα όλα αυτά τα θέματα να τα αφήσουμε ως έχουν, ως αντικείμενο δηλαδή, ακριβώς αυτό αυτών των διαβουλεύσεων που θα πρέπει να διεξαχθούν στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο με την υποστήριξη και συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό το πλαίσιο και του Τζέραλντ την τροπολογία που αναφέρεται ότι για το 2005 που θα πρέπει να ε, αναφέρεται στο θέμα αυτό και πρόκειται για μια απλή τροπολογία, ωστόσο όμως ε, δεν νομίζω ότι συμβαίνει απόλυτα αυτό και τεχνικά και για νομικούς λόγους. Επίσης και επειδή δεν πρόκειται να ενδυναμώσει την πολιτική συνένεση, δεν θα την τονώσει όσον αφορά τις ε, την διακομματική συνένεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων του Κοινοβουλίου και προσπαθώ να δημιουργηθεί αυτή η υποστήριξη για τις θεμελιώδεις προτάσεις, ε, θεμελιώδους σημασίας ε, όσον αφορά την ε, συνταγματική αυτή πτυχή. Και ξέρουμε ότι η Κροατία έχει αυτή την ε, εκκρεμότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα υποβληθεί μια πρόταση για την ε, ανακατανομή των ε, εδρών έγκαιρα για τις εκλογές του 2014. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπερβάλλουμε σήμερα επ' Καθώς αντιμετωπίζουμε την προοπτική μιας συντακτικής συνέλευσης ως προοπτική είναι σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο να είναι απόλυτα προετοιμασμένο με έναν συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο με ένα πακέτο εκλογικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά το εκλογικό δίκαιο ώστε έγκαιρα όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν αυτές οι εκλογές και να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτών των αρχών να είμαστε έτοιμοι. Θα ήθελα να μπορέσουμε το Δεκέμβριο να εγκρίνουμε, να ψηφίσουμε προς έγκριση ή τον Ιανουάριο το αργότερο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε μέχρι τότε να έχουμε αποσαφηνίσει το σενάριο της διακυβερνητικής διάσκεψης ή της συντακτικής συνέλευσης μέσα στο διακυβερνητικό πακέτο προτάσεων και όλων των άλλων θεμάτων που θα πρέπει να γίνουν ώστε να ενδυναμωθεί η νομιμοποίηση, η πολιτική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή να είναι σαφέστερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γουαλτιέρη. Έχει ζητήσει το λόγο. θα προτιμούσα να ακούσω πρώτα την άποψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γιατί η κατάσταση έτσι όπως παρουσιάζεται είναι γνωστή και η άποψη της ομάδας μας είναι σαφής. Εμείς υποστηρίζουμε την πρώτη διατύπωση της έκθεσης. Συμφωνούμε με τη βασική ιδέα του εισηγητή να παρουσιάσει ε, μια θα έλεγα διαφορετική βερσιόν η οποία δίνει περισσότερα περιθώρια διαπραγματευτικά και προς το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά οι θέσεις μας δεν αλλάζουν και μένουμε στις συζητήσεις που είχαμε κάνει στο παρελθόν. Αυτό το οποίο κάνει τη συζήτηση λοιπόν περίπλοκη είναι οι θέσει των υπολείπων πολιτικών ομάδων. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο λοιπόν εδώ, να επαναλάβω ότι η θέση μας να επαναλάβω ίσως τους λόγους για τους οποίους ε, θεωρούμε και μένουμε ότι η έκθεση πρέπει να γίνει δεκτή από την Ολομέλεια. Παράλληλα νομίζω ότι η πρόταση του εισηγητή να παρουσιάσει μια διαφορετική, πιο ευέλικτη διατύπωση εμένοντας και στις ε, συνδέσεις ανάμεσα στην έκθεση αυτή με τις μελλοντικές αλλαγές της συνθήκης είναι μια σοφή πρόταση γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει το θέμα της α, συντακτικής συνέλευσης, της διακυβερνητικής με, περιορισμένα, α, με περιορισμένες αρμοδιότητες κτλ. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να δεσμευτούμε ιδιαίτερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν είναι καθόλου λάθος σαν αντίληψη και νομίζω ότι η συγκεκριμένη αυτή τροπολογία δεν είναι τελικά απαραίτητη. Απλά μας δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε τα προβλήματα της κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αφήσουμε για να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο μέλλον και αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει δεκτό από το Κοινοβούλιο και τη συγκεκριμένη Επιτροπή, τη δική μας δηλαδή. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συνεχίσουμε όπως ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε και στο παρελθόν και περιμένουμε τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επ' αυτού. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σχολιάσετε λίγο αυτά τα οποία ζητώ. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Σέπλεν έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα αυτά, αλλά νομίζω έχει επέρθει κάποια κόπωση. Συζητούμε αυτό το θέμα πάρα πολύ καιρό. Δεν σημαίνει ότι είναι σήμαντο ή ε, λεπτομέρεια, αλλά γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες και τα επιχειρήματα. Βέβαια, ε, τα πράγματα άλλαξαν αλλού στην παγκόσμια κατάσταση. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν. Είναι θέμα όμως νομιμότητας, καταλαβαίνετε. Είναι απολύτως κομβικό και κρίσιμο. Σε ό,τι αφορά το πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο, γιατί αυτό μας απασχολεί, ε, είναι σαφές ότι το κοινοβούλιο είναι διχασμένο σε αυτό το θέμα και οι διάφορες πολιτικές ομάδες αν δείτε τι τροπολογίε. αυτό αντανακλούν και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα έντονο. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ΕΛΚ δεν έχει ενιαία θέση αποκρισταλωμένη. Άλλα μέλη έχουν μια άποψη ε, πολύ ισχυρή άλλοι λιγότερο, γιατί εδώ που κατά πόσο είναι απαραίτητο ένα πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Όλα έχουν να κάνουν με την ομαλή λειτουργία, ε, το πώς ρέουν τα πράγματα σε αυτό το ρευστό κόσμο που ζούμε. Η αρχή είναι καλή, είναι απαραίτητη. Είναι πολλά τα θέματα που μας απασχολούν, αλλά η ερώτηση που είναι και πάλι ρητορική ίσως, αλλά ε, με ουσιαστικό νόημα. Είναι τώρα καιρός για τέτοια πράγματα. Είναι του παρόντος, δεν είμαι πεπισμένος. Γιατί αν ε, δεν είναι του παρόντος δεν θα βρει και την υποστήριξη που αξίζει. Από όσα διαβάζω, ε, έχω ξεκάθαρο εγώ στο μυαλό μου ότι αυτή η υπόθεση έχει πολύ λίγη υποστήριξη εκτός του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ το υποστηρίζω το πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Αλλά πέρα από το θέμα της νομιμότητας, ε, είναι και το ζήτημα αν υπάρχει πραγματικά ένας ευρωπαϊκός λαός, Δήμος, με την αρχαιολινική έννοια. Και για την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι πραγματικά κρίσιμο θέμα εδώ και κλειδί Και αυτό που θα συμβεί, μάλλον ήδη συμβαίνει, είναι κάποια συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών. Που αυτό σημαίνει απαραίτητα συγκέντρωση της εξουσίας, που δεν θα έχει πανευρωπαϊκή αντιπροσώπευση ή εκπροσώπηση. Εγώ μπορεί να έχω μια καταφατική απάντηση, αλλά πολλοί δεν έχουν πιστεί ακόμα. Αν γίνει συντακτική συνέλευση και μάλλον προς τα εκεί πηγαίνουν τα πράγματα με επόμενη διακυβερνητική διάσκεψη θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα είναι μόνο για την οικονομική διακυβέρνηση ή και για την εκλογική διαδικασία. Εγώ θα έλεγα το δεύτερο μάλλον, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Χρειάζεται συζήτηση και η θέση μου είναι από τη μια να το υποστηρίζω, αλλά πρέπει να συζητήσω και με την ομάδα μου και να λάβω υπόψη ε, και τις ε, άλλες φωνές της ομάδας. Κύριο έχει δει το λόγο. Η πρόταση να έχουμε αυτού του 25 ευρωβουλευτέ που θα εκλέγονται σε πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο είναι μια μετροπαθής ε, σε σχέση με τις ε, πανευρωπαϊκές τάσεις ε, για εκείνους που βρίσκονται εκτός όμως θέτει κάποια ερωτήματα αν έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες ευρωβουλευτών που θα εκλέγονται με δύο διαφορετικά συστήματα ποιο θα είναι το ανώτερο σύστημα και το ε, υποδέστερο αν η πανευρωπαϊκή λίστα θα είναι το προτιμόμενο θέμα, γιατί να περιοριστούν σε 25 αυτοί οι ευρωβουλευτέ. Αν δει κανεί τις τροπολογίες, η τροπολογία 21 θέλει να έχει 10% του συνολικού αριθμού, 75. Αν όχι, αν, τότε 75 γιατί όχι 751. Και αυτό απηχείται εδώ. Δεν θα ήταν αυτός ο στόχος τελικά όχι υποχρεωτικά ημών αλλά άλλων να είναι όλο το κοινοβουλίο που θα εκλέγεται με ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο εκλογές τώρα σε ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο ευνοούν κόμματα που έχουν μια πλήρως δεσμευμένη ε, φιλευρωπαϊκή προοπτική και πέρα από αυτό με απήχηση σε εκείνους ε, από τους πολίτες που θα έχουν κίνητρο να πάνε να ψηφίσουν αυτούς τους ευρωβουλευτές γιατί διαφορετικά θα βρουν αυτό τον πίνακα ε, ότι δημιουργεί αυτή η πανευρωπαϊκή λίστα ή σύγχυση ή δημιουργεί προβλήματα. Ευχαριστώ. Ho ascoltato la sua premessa. Άκουσα την εισαγωγή σα είπατε ότι το θέμα αυτή το συζητάμε εδώ και χρόνια όπω και τον κώδικα συμπεριφορά των κοινοβουλευτικών. Δεν θα ήθελα να βοηθήσω και εγώ στο να μακρηγορούμε στη συζήτηση αυτή, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία την οποία έχει ξεκινήσει η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω μια όχι απλά γενική θετική αξιολόγηση αυτού του ευρωπαϊκού ψηφοδελτίου και θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα. Γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι συνάδελφοι ότι υπάρχει ένα αδυσεπίλητο πρόβλημα στο κοινοβούλιο αυτό. Για την νομοθετική περίοδο 90 με 2004 και για τα προνόμια των βουλευτών είχε εγκριθεί μία πρόταση σχετικά με τον κανονισμό των βουλευτών με πολύ μεγάλη πλειοψηφία για όλη αυτή την περίοδο σχετικά με την ασυλία και τις εγγυήσει για τον Ευρωβουλευτή ε, που είναι κάτι το οποίο είναι υπεράνω της αναφοράς των ισχυόντων στα διάφορα κράτη-μέλη. Στα διάφορα κράτη-μέλη βέβαια ισχύουν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την ασυλία αυτή. Εμείς ε, εγκρίναμε εκ νέου την βασική αυτή ιδέα όταν προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε τα θέματα τα οποία αφορούν τα πρακτικά προβλήματα των βουλευτών όπως οι αποζημιώσεις κτλ. Και το 2009 ψηφίσαμε πάνω σε αυτό με ισχυρή πλειοψηφία. Γιατί να μην κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια και μιας και υπάρχουν οι τροπολογίες Γκουαλτιέρη σχετικά θετικές, νομίζω το να δούμε ακριβώς τι εγγυήσει μπορούμε να δώσουμε προς την λειτουργία του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να μην περιμένουμε δηλαδή συζητήσεις ε, σε βάθος με το Συμβουλίο, αλλά να κάνουμε μία πρόταση η οποία να περιλαμβάνει αυτό το οποίο ανήκει στην ε, συνθήκη ε, ή μάλλον στον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που δεν, έγινε, δεν ελήφθη υπόψη διότι το Συμβούλιο προχώρησε σε μια εντελώς διαφορετική και μεγαλύτερη σε μέγεθος ρύθμιση εκ των υστέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό αυτό το θέμα. Πού είναι ε, εδώ η στρέβλωση. Όχι ότι δεν υπάρχει ενθουσιασμός ε, που είπε ο κύριος Σέφλιν, αλλά είναι ότι δεν υπάρχει κυριος σεφλιν αλλα οτι προοπτική για αυτή την πρόταση για να εγκριθεί ε, από το Συμβούλιο. Εμείς έχουμε περιορισμένο χρόνο για αυτό το θέμα και είναι κεντρικό να ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα. Γιατί είμαστε αντίθετοι με αυτό το θέμα. Κάθε βήμα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση δημιουργεί θεσμικά όργανα χωρίς καμία συμμετοχή του κοινού, για να μην πω ενθουσιασμό. Ο κύριος Σόφλη είπε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός, ε, δεν έχουμε Δήμο. Έχουμε κράτος όμως, χωρίς Δήμο. Δηλαδή δημιουργούμε θεσμικά όργανα, δημιουργούμε κράτος, θεσμούς πολιτιακούς, χωρίς να έχουμε Δήμο. Ε, υποστήριξη, δημοκρατική νομιμότητα για να δικαιολογούν την ύπαρξη των θεσμικών μας οργάνων. Με τη θεωρία ότι καλά θα ακολουθήσει η κοινή γνώμη. Αυτό όμως δεν μας βγαίνει ως θεωρία από την πράξη. Κοιτάξτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού. Από το 79 μέχρι το 94 ε, και μέχρι σήμερα πέφτει συνέχεια. Ε, ε, εγώ εξελέγη με συμμετοχή 24% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότεροι ψήφισαν την επομένη για το Big Brother, για το ποιος θα βγει από το σπίτι έχει πέσει πάρα πολύ ε, ε, η συμμετοχή και η δημοτικότητα ε, και μέχρι το 2009. Τη θεωρία λοιπόν την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δοκιμάσει ότι αν δεν είναι κανείς περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει κοινή γνώμη. Όχι. Τα στοιχεία σήμερα αποδεικνύουν το αντίθετο. Κανένας ενθουσιασμός πουθενά. Ούτε στην εκλογική μου περιφέρεια, ούτε πουθενά σε κανένα κράτος μέλος για να προχωρήσουμε έτσι προς ένα πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο. Λες και είμαστε ενιαία περιφέρεια. Για το λόγο αυτό η ομάδα μου θα το καταψηφίσει. Ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κάποιες πατρίες προς τον συνάδελφο σε σχέση με την συμμετοχή στις εκλογές ε, όπου αναφέρθηκε αν έχουμε γενικές ε, τέτοιες συγκρίσεις όσον αφορά τις ευρωεκλογές ε, θα έλεγα ότι αυτό δεν θα ήταν θεμητό διότι το 2004-2009 και προηγούμενα ήδη μπήκαν νέα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παραδοσιακά είχαν πολύ χαμηλότερη συμμετοχή ακόμα και στις εθνικές τους εκλογές και γι' αυτό πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε ποιο είναι, ποιος είναι ο μέσος όρος των συγκρίσιμων χωρών σε σχέση με τις ευρωεκλογές ίσως μπορεί να είναι χαμηλότερο αλλά πάλι είναι συγκρίσιμο σε σχέση με τη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές. Στην Γερμανία το 2009 είχαμε για πρώτη φορά συμμετοχή ψηλότερη από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα, σε σχέση με τις προτάσεις που έχουμε στο τραπέζι, ρητά παραπονούμε για το ότι για τις 25 επιπλέον αυτές έδρες έχουμε αντιπαράθεση και δημιουργούμε τριβές. Νομίζω ότι παρακάμπτουμε έτσι, αγνοούμε την εντολή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Για τις 25 ε, αυτές έδρες ε, είναι ίσως μια καλή ιδέα. Διαρωτώ με γιατί να είναι 25 αυτοί που θα εκλέγονται και γιατί όχι 43, γιατί όχι 17 αν και το λογικότερο θα ήταν να έχουμε έναν αριθμό που να ανταποκρίνεται στον αριθμό των κρατών μελών, ώστε θεωρητικά να μπορούσαμε να πετύχουμε με αυτή την πανευρωπαϊκή λίστα να μπορούν να εκλέγονται από κάθε κράτος ε, ευρωβουλευτές αν θα το ήθελαν έτσι οι ε, εκλογείς αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν βρίσκονται στις συνθήκες ε, και για το, ε, τα όσα κυοφορούν εδώ και πολύ χρονικό διάστημα θα έπρεπε να δούμε πώς είναι δυνατόν στην εφαρμογή να ε, υλοποιηθούν. Αλλά εκεί όπου η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέτει γνώμονα και θέτει τον πύχη για αυτά τα πράγματα, εδώ όμως πρέπει να δούμε ότι είναι το άρθρο 14 και το ε, άρθρο για την, ε, ε, τις διαδικασίες γίνεται λόγος για το εκλογικό δίκαιο και είναι δυσκολότερα τα πράγματα διότι για κάποια τροποποίηση απαιτείται τροποποίηση της συνθήκης. Για το 2014 γίνεται σαφής λόγος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει μια πρόταση και αυτή την πρόταση δεν την κάνουμε τώρα εμείς. Γι' αυτό έλαβα την ελευθερία με την τροπολογία αυτή σε σχέση με το 27 με τη δική μου πρόταση να έχουμε σαφή ρύθμιση πώς αυτές οι 751 έδρες θα συντίθενται πώς θα προβαίνουμε στη σύνθεση αυτή και θα υποβάλω αυτά τα στοιχεία στους συναδέφους. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η πρώτη παύλα της τροπολογίας 27 ίσως ε, ε, αφορά κάποιο γλωσσικό σφάλμα τουλάχιστον στα αγγλικά διότι γίνεται λόγος για εκλογικές περιφέρειες και στη δική μου διατύπωση στα γερμανικά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θέλω να έχουμε μια σαφή ρύθμιση, να έχουμε ένα κανόνα που θα λέει 75% 75% που θα μπορεί να επεξηγηθεί όσον αφορά ε, τους ε, ε, πολίτες γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κατανόηση για τέτοια θέματα όπως εκλογική συμμετοχή σε εκλογές εκπροσώπηση και το Cambridge Compromise και άλλες διατυπώσεις που έχουμε αν εδώ έχουμε προσκαλούμε καθηγητές μαθηματικών και δεν καταλήγουμε στο με δέκα προτάσεις ε, να μπορέσουν να επεξηγήσουν ε, την ε, προσέγγιση τους, τότε δεν είναι χρήσιμη η δική τους προσέγγιση και είναι για τον κάλαθο των αχρήστων. Επιτρέψτε μου συνάδελφε Ντάφ. Ομολογώ ότι πρόκειται για ένα γερμανικό, ας το πούμε, μια γερμανική προσέγγιση και γερμανικό θέμα, αλλά είναι και θέμα άλλων κρατών μελών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διοργανωτική προσέγγιση ε, λογικού χαρακτήρα και η πρόταση ε, θα αναφέρεται σε ένα ποσοστό ε, ενιαίο και μετά η αρχή DONT για την αναλογική εκπροσώπηση όπου ένα μέρος των ψήφων θα σταθμίζεται και ανάλογα με τον πληθυσμιακό ε, το πληθυσμιακό εύρος ε, των διαφορετικών χωρών θα έχουμε την διαφορετική εκπροσώπηση. Και εδώ σε σχέση και με την άσκηση προσφυγής ε, σε συνταγματικά δικαστήρια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυσκολίες στις εθνικές κυβερνήσεις αν δεν υπάρξουν σαφείς ρυθμίσεις, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε με τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια σε μια λειτουργική προσέγγιση και σε μια ας το πω έτσι ίσου, ίσου προς να αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι κατανοώ τα επιχειρήματα του κυρίου Νταφ. Είναι πολύ σωστά προπαρασκευασμένα, αλλά παρόλα αυτά οφείλω να πω ότι δεν θεωρώ ότι έχει φτάσει ο καιρός για να περάσουμε σε μια τέτοια φάση. Θα πρέπει να περιμένουμε έτσι ώστε τα κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν γνωστότερα σε εθνικό επίπεδο. Αν είχαμε εκλογές τέτοιου είδους ε, σύντομα, διαρωτώ με αν όλα τα μέλη μας θα εγνώριζαν ε. Ε, πριν εκλεγούμε σε ποιο κόμμα θα ήμασταν. Θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική, δεν είμαι σίγουρος για αύξηση στην εκλογική προσέλευση, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος. Και να πω επίσης ότι σαν παράδειγμα πέρυσι ή και φέτος όταν στην Φιλανδία κάναμε τις εκλογές μας, η ευρωπαϊκή διάσταση ήταν ένα μόνο από τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση. Και παρόλα αυτά η συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι άλλες εποχές. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ήταν ικανοποιημένος ο κόσμος, αλλά σίγουρα η διαδικασία ήταν δημοκρατική. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα, θα έλεγα, πραξικόπημα επίσης των μεγάλων κρατών μελών, γιατί όταν χρησιμοποιούμε το σύστημα default οι υποψήφοι θα προέλθουν από ό,τι φαίνεται πρώτα από τις μεγάλες χώρες και αυτοί θα έχουν τις περισσότερες αρμοδιότητες αλλά αν πράγματι θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή θα πρέπει να, ελέγξουμε, ε, να επιλέξουμε συγγνώμη, υποψηφίους οι οποίοι να είναι πανευρωπαϊκώς γνωστοί. Από ό,τι όμως φαίνεται εδώ δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα τα οποία να είναι γνωστοί σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο Άρη Βάτανεν θα μου πείτε. Πράγματι ο Άρη Βάτανεν θα μπορούσε να πάρει μια έδρα η Φιλανδία. Ήταν ένας πολύ καλός επίσης βουλευτής και τον εκτιμώ, αλλά δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουμε να επιλέξουμε τραγουδιστές, ηθοποιούς και τέτοιου είδους ανθρώπους που είναι οι μόνοι γνωστοί ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Αγγέλα Μέρκελ βέβαια θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο πρόσωπο γιατί είναι πάντα στην επικαιρότητα και όλοι οι πολίτες μας γνωρίζουν ποια είναι η συγκεκριμένη κυρία. Αλλά η επιλογή θα είναι θα έλεγα ανάμεσα σε ονόματα τα οποία δεν είναι εδώ και δεν εργάζονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό ενώ θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο. Λοιπόν, δεν έχει φτάσει ακόμα η κατάλληλη στιγμή λοιπόν και πρέπει να περιμένουμε mm. πριν δεχτούμε μια τέτοια πρόταση. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, υπάρχουν ε, πάρα πολλοί οι οποίοι είναι κατά. Η δική μου ομάδα δεν έχει συγκεκριμένη άποψη ακόμα διαμορφώσει και ίσως να μην μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση αυτή την οποία εγώ δεν δέχομαι ah, Λοιπόν Αλλά πρώτα ο κύριος Μέντες δεν Κύριε Πρόεδρε πιθανότατα ίσως η καλύτερη απόδειξη ότι δεν έχει οριμάσει το θέμα είναι ότι οι συνάδελφοι που τους εκτιμώ βαθύτατα και ξέρω ότι είναι ευρωπαϊστές συζητούν ακόμα με εθνικότητες ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα Φιλανδό, ένα Τσέχο, ένα Ισπανό. Μα δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Τι να βάλουμε 27 για να χωράει ένας από κάθε εθνικότητα. Ε, τότε δεν έχουμε χαπάρι πάρει. Πρόκειται για την ιδεολογία ε, τις αξίες και τις αρχές των ευρωπαϊκών κομμάτων και δεν έχει σημασία ούτε η εθνικότητα ούτε το μέγεθος της χώρας. Αν ακόμα σκεφτόμαστε με τέτοιους χώρους που θα χωρέσει ο Μαλτέζος και ο Σλοβάκος, χαιρετίσματα. Είναι απογοητευτικά αυτά κύριε Πρόεδρε. Και ζητώ συγγνώμη έτσι που εξεράγει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λοιπόν, θα προσπαθήσω όσο μπορώ και εγώ να συνεισφέρω στη συζήτηση. Πρώτον, είναι σαφές ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αποδίδει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την δυνατότητα να διατυπώσει πρόταση μετά από δική του πρωτοβουλία για ενιαίο εκλογικό νόμο. Αυτό είναι σαφές. Είναι σαφές επίσης ότι ένας τέτοιος νόμος θα ήταν ένα πολύ ισχυρό σύμβολο και τα σύμβολα δεν είναι πάντα άχρηστα θα έλεγα. Είναι ένα ισχυρότατο σύμβολο προόδου θα έλεγα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν σε σχέση με αυτό και γι' αυτό σαν βουλευτής και σαν πρόεδρος της Επιτροπής εγώ συμφώνησα με την ιδέα να προσπαθήσουμε να εγκρίνουμε τον ενιαίο εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής περίοδου. Αλλά απερίφθη η πρόταση αυτή στην πρώτη φάση και η απόρριψη αυτή οφείλεται σε μια πραγματική διαίρεση της γνώμης στο εσωτερικό των κομμάτων. Δεν νομίζω ότι η σοσιαλιστική ομάδα είναι συμπαγής υποστηρίζοντας την πρόταση Νταφ. Και το ίδιο όπως είπε και η προλαλήσασα για τη δική της ομάδα, τους φιλελευθέρους. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προχωρήσουμε ή θα πρέπει να παρετηθούμε από την προσπάθεια σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Αν θέλουμε για μια ακόμη φορά να κατεβούμε στην Ολομέλεια και για μια ακόμη φορά να απορριφθεί η πρότασή μας, δεν ξέρω τι νόημα έχει κάτι τέτοιο. Το θέμα λοιπόν το οποίο τίθεται σε αυτή τη φάση είναι το θέμα του ενιαίου εκλογικού ε, χώρου Ευρωπαϊκού Εκλογικού Χώρου. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία είναι αντικείμενο απορίας και συζήτηση σε αυτή τη φάση. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επίλυση κάποιων από τα προβλήματα αυτά. Μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σαφέστατο κριτήριο για την κατανομή των εδρών. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Ας καταλήξουμε αν είναι δυνατόν σε ένα αυτόματης εφαρμογής κριτήριο για την κατανομή των εδρών. Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες, έγινε και το σεμινάριο στο Κέμπριτζ, έγιναν προτάσεις και δεν είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι θέλει ο κόσμος. Κατανοώ επίσης ότι η παρουσία των κρατών μελών και η παρουσία τους και στο Κοινοβούλιο με την ταυτότητά τους είναι κάτι το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο βάρος και δεν προσμετράται μόνο από την ποσόστοση της κάθε χώρας στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου αυτή η εικόνα θα έλεγα. και αν πάρουμε κάποιες αποφάσεις σχετικά με τη συμπίεση σαν παράδειγμα των εδρών άνω των 91 που μπορεί να έχουν κάποιες μεγάλες χώρες ε, ή το αντίθετο για τις χώρες που έχουν κάτω από 91 προφανώς αυτά είναι θέματα που μένει ακόμα να συζητηθούν είναι ένα πρόβλημα, είναι μια εκκρεμότητα. Η πρόταση Γκαργκάνη θα έλεγα για τις αποζημιώσεις και τα πλεονεκτήματα και την ασυλία σίγουρα δεν είναι μια κακή ιδέα. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον εκλογικό νόμο. Είναι μια πρόταση μεταρρύθμισης αν θέλετε του ισχύοντος καθεστώτος. Ναι, έχουν κατατεθεί και τροπολογίες λέει ο κύριος Γκαργκάνιε. Αλλά παρόλα αυτά Αυτά, εν πάση περιπτώσει, είχα να πω. να πω ότι δεν πρέπει να πάρουμε απόφαση σε αυτή τη φάση να μην κάνουμε τίποτα αλλά ας μην πάρουμε και την απόφαση να πάμε και να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο σε μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια της οποίας γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Ίσως ακόμα και σήμερα ή την επόμενη φορά σε επίπεδο συντονιστών να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κάποια λύση Έχω αμφιβολίες ε, αν μπορούμε να βρούμε μια τέτοια λύση, αλλά ας προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Νταφ. Ο κύριος Γαργάνη έχει ζητήσει το λόγο. Είχα την αίσθηση ακούγοντας τη συζήτηση αυτή και είναι ένα θέμα θυμίζω το οποίο γνωρίζω εδώ και αιώνες θα έλεγα θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο μας διαιρεί είναι ο εθνικός εκλογικός κατάλογος, η εθνική εκλογική λίστα. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Η ευχή για ένα ενιαίο εκλογικό σύστημα, που είναι μια ευχή η οποία έχει ακουστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει οριμάσει ακόμα. Εφόσον υπάρχουν διαιρέσεις βέβαια στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων, φοβάμαι ότι θα προκαλέσει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Δεν μπορούμε όμως όλα τα υπόλοιπα να προσπαθήσουμε να τα ξεχάσουμε ή να τα πετάξουμε στη θάλασσα όλα τα θέματα τα επιμέρους έχουν θα έλεγα μια κάποια σημασία και όλα αυτά μαζί είναι εγγυήσει για την κατάλληλη εκπροσώπηση των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει λόγω των δυσκολιών οι οποίες υπάρχουν να απορρίψουμε όλες τις προτάσεις οι οποίες ε, ε, ε, οι οποίες σε αυτή τη φάση μας διαιρούν, σε αυτή τη φάση μας διαιρούν. Ο λαός της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες, έχει εκφραστεί. Ε, κάποιες χώρες ψήφισαν με πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχή. Στη Ρουμανία ήταν 29% αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να κάνει μια πρόταση πάντως στο Κοινοβούλιο. Αυτό δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Να σχολιάσω και εγώ τα τελευταία που ακούστηκαν και το τι πρέπει να γίνει, λέει ο κύριος Γκουαλτιέρη. Δεν νομίζω ότι το θέμα της υπερεθνικής αυτής λίστας εκλογικής είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Εγώ νομίζω προσωπικά, όπως και ο κύριος Νταφ, ε, έχουμε κάποιες προτάσεις κάνει. Αν ο κύριος Γκαργκάνη μπορεί να κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, εμείς θα τις εξετάσουμε με το μέγιστο δυνατό ενδιαφέρον. Πάντως, το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουμε σε σχέση με τη βασική πρόταση την οποία κάνει η έκθεση του κυρίου Νταφ. Στην πραγματικότητα, Πρόεδρε, είναι ότι η έκθεση αυτή δεν έγινε δεκτή με μία ψήφο διαφορά στην Ολομέλεια αποφασίστηκε να μην ψηφιστεί καν γιατί υπήρχαν θα έλεγα αμφιβολίες για τη διαμόρφωση μιας ικανής πλειοψηφίας. Ήταν μια σοφή απόφαση για να μην χάσουμε χρόνο. Και στη συζήτηση που κάνουμε σήμερα δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε τη διαδικασία από εδώ και πέρα σωστά. Πάντω, ένα περιορισμένο χρόνο χρόνος, δύο-τριών εβδομάδων, ενό μηνός που θα επιτρέψει στι πολιτικές ομάδες να κάνουν τι εσωτερικές τους και ε, ε, θα έλεγα ενέργειε για να καταλάβουν πού μπορούν να καταλήξουν, είναι κάτι που θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε ένα επιχείρημα που θεωρώ αποφασιστικό. Μιας και έχει αλλάξει το σκηνικό από ότι τους τελευταίους μήνες το θέμα μιας ισχυρής οικονομικής ένωσης και η υπεραιτέρω ολοκλήρωση και η υπεραιτέρω αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οικονομικά θέματα είναι υποσυζήτηση. Αν αυτή η πρόταση ακολουθηθεί και από την ενίσχυση του συστήματος νομιμοποίησης δημοκρατικής της προσπάθειας αυτής ολοκλήρωσης, τότε η προσπάθεια θα γίνει καλύτερα κατανοητή και από συναδέλφους και από εθνικές συνιστώσεις οι οποίες εδώ και λίγους μήνες έχουν δείξει ότι είναι ιδιαίτερα διστακτικές. Πέραν λοιπόν αυτού του εσωτερικού ελέγχου που μπορούν να κάνουν οι πολιτικές ομάδες θα αποφασίσουμε ανάλογα με το αποτέλεσμα της το τι θα κάνουμε αν θα περάσουμε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια και πότε. Θα πρέπει να ελέγξουμε, να δούμε αν οι πολιτικές ομάδες θα στηρίξουν μια ψηφοφορία στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια να δούμε αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις πολιτικές. Λοιπόν, ο κύριος Νταφ πρέπει να απαντήσει, έχουν ακουστεί πολλές απόψεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γκουαλτιέρη και τον κύριο Μέντες Δεβίγκο για την υποστήριξή τους. Σημερίζομαι ε, την αυξανόμενη απογοήτευση που νιώθω. Ευχαριστώ και τον κύριο Σέφλιν για την υποστήριξή του. Γνωρίζει ότι δεν συμφωνώ με αυτή τη θεωρία του Δήμου του ευρωπαϊκού ε, λαού, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό ούτε επιθυμητό στο κάτω-κάτω να έχουμε ένα λαό ευρωπαϊκό πριν αποκτήσουμε πλήρη ε, ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη η οποία να εμπνέεται και να καθοδηγείται από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε ε, ομοσπονδιακό επίπεδο. Και αυτό θα έχει νόημα για τα ευρωπαϊκά ζητήματα που μας απασχολούν εδώ στο Κοινοβούλιο. για να ασχολούμαστε με τρόπο συνεχή και ομαλό, με μόνιμη επαφή με το εκλογικό σώμα. Αλλάζει και η ποιότητα της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής και θα αυξηθεί και η υποστήριξη. Σέβομαι και τιμώ την Ανελή Τεμάκη, αλλά ε, όλοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι τα εθνικά κόμματα και οι εθνικοί υποψήφοι είναι πιο κατάλληλοι για ευρωπαϊκή εκπροσώπηση και εκλογή, νομίζω υπερβάλλουν. Έχουμε δει και στο παρελθόν τα εθνικά κόμματα πώς φιλοδοξούν να δρουν ε, αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και από αυτό νομίζω πορεύει και εξηγείται το πρόβλημα της χαμηλής συμμετοχής ε, στις ευρωεκλογέ. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Και το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης τώρα ή της μεγαλύτερης φορολογικής ενοποίησης θα χρειαστεί και πιο ομοσπονδιακού τύπου διακυβέρνηση και αυτό ακριβώς είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να βρούμε έναν τρόπο να αντικατοπτρίζεται η ανάγκη ε, της δημοσιονομικής αλληλεγγύης όχι μόνο μεταξύ κυβερνήσεων και φορολογημένων αλλά και μεταξύ ε, ψηφοφόρων. Καλωσορίζω και την παρουσία του κυρίου Γκαργκάνη για διάφορους λόγους και προσωπικούς και επίσης γιατί ξέρω ότι εκτιμάει τη σημασία των θεμάτων ε, ασυλιών και προνομίων. Κατέθεσα μια βελτιωμένη νέα έκδοση των προτάσεων του Κοινοβουλίου από το 2005 για να αναθεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο το οποίο είναι παράτημα της έκθεσής μου. Απαντώ στον κύριο Μπρόνς ότι δεν προτείνουμε διάφορες κατηγορίες ευρωβουλευτών. Αυτή τη στιγμή εκλεγεί ο κάθε ευρωβουλευτής θα είναι ε, ίδια η εντολή όλων. Αλλά θα έρχονται εδώ με διαφορετικούς τρόπους, όπως εκλέγονται και σήμερα με διαφορετικούς τρόπους. Οι εκλογικέ διαδικασίε, τα εκλογικά συστήματα στα διάφορα κράτη-μέλη είναι μέχρι και αντιβατικά μεταξύ του. Και δεν νομίζω ότι αυτό προσθέτει κάτι στην ε, περιπλοκότητα, την ήδη υπάρχουσα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Ούτε μπορώ να μιλήσω για τις μελλοντικές γενναίες. είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα να μιλάει κανείς εξ ονόματος παρούσης επιτροπής σήμερα. Χωρίς να προεξοφλώ, να προβλέπω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Διαδικασία. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ε, ε, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα στην Επιτροπή μας Αυτό θα καθοδηγήσει καλύτερα τις πολιτικές ομάδες, μια ε, σαφής κατεύθυνση που θα δώσει η Επιτροπή μας, θα τους βοηθήσει. Και σε σχέση με τα όσα είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιμείνω να ψηφίσουμε ενδεχομένω τον Ιανουάριο εδώ στην Επιτροπή και στη διαδικασία αυτή θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και μερικά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή σας ανησυχούν. για το θέμα της αναλογικότητας προοδευτικά μειούμενης και το πώς κατανέμονται οι έδρες με βάση μαθηματικούς τύπους. Όλα αυτά θα βρεθούν μόνο μέσα από διάλογο με το Συμβούλιο. Ο κύριος Βίλαντ ε, αναγκάστηκε να φύγει και ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Αν ήταν παρόν όμως θα το απαντούσα λέγοντας ότι το αποτέλεσμα της ε, δικής του πρότασης στη δροπολογία 27 είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που θα έβγαινε από τη διαδικασία του συμβασμού του Κέμπριτζ. Λοιπόν, ας πάρουμε τώρα μια βαθιά αναπνοή και ας προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο που έχουμε χαράξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάναμε μια, για μια ακόμη φορά μεγάλη συζήτηση. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σε επίπεδο μεθοδολογίας. Κάποιοι είπαν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων. Να μην ορίσουμε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών και ε, συζήτηση. Άλλοι πιστεύουν ότι έχουμε συζητήσει επί μακρό, να περάσουμε σε ψηφοφορία, οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο, από ό,τι φαίνεται, 26 Ιανουαρίου. Οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί Κάποιες έχουν γίνει ήδη αντικείμενο συζήτησης, όχι συνολικά βέβαια, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες επιλογές. Αυτό που είπα εγώ δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ημερομηνία για ψηφοφορία. Μπορούμε να βάλουμε τις 16 Ιανουαρίου αν θέλετε, 26 δεν ξέρω. Κοιτάξτε εγώ θα προτιμούσα να δω αν υπάρχει μια κάποια ευρύτερη συνένεση πρώτο να μην ορίσουμε την ημερομηνία για ψηφοφορία στην Επιτροπή, έτσι ώστε τις επόμενες εβδομάδες οι πολιτικές ομάδες να καταλήξουν κάπου για τη θέση τους. Η άλλη λύση είναι ότι υπάρχουν οι τροπολογίες, οπότε βάζουμε συζήτηση στις 26 Ιανουαρίου. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της του να ορίσουμε, να κάνω μια τρίτη πρόταση, λέει ο κύριος Γκαργάνη. για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τις υπάρχουσες τροπολογίες. Μπορούμε να καταθέσουμε μια νέα προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, μια επιπλέον προθεσμία. Ο κύριος Νταφ. Κοιτάξτε, θέλετε να ψηφίσουμε και αυτή την πρόταση του κύριου Γκαργάνη. Θα ήθελα, ναι. Με κάθε σεβασμό όμως πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί, τα θέματα έχουν συζητηθεί επί πολλούς μήνες πλέον και αυτό που χρειάζεται είναι να πάμε στις κοινοβουλευτικές ομάδες με μια σαφή θέση αυτής της κοινοβουλευτικής επιτροπής που πρέπει να αποκρισταλωθεί. Γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε την διαδικασία τροπολογιών και να περάσουμε στην ψήφιση προς έγκριση στις 27 Ιανουαρίου. Νομίζω αυτό θα έπρεπε να γίνει. Αναμένει το Κοινοβουλίο να συμβεί αυτό, να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Η καθυστέρηση όσον αφορά την κατανομή των εδρών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ήταν ούτως ή άλλως ε, ως καθυστέρηση και λόγω του θέματος της Κροατίας θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα πρέπει να συμφωνήσετε ή όχι. Πότε θέλετε να ψηφίσουμε με τις προθεσμίες οι οποίες προτάθηκαν για την 26η Ιανουαρίου. Ποιοι θέλουν ψηφοφορίες 26 Ιανουαρίου. 7, 8. Ποιοι θέλουν να περιμένουμε ακόμα περισσότερο και να συζητήσουμε μέσω των συντονιστών το πότε θα γίνει η νέα ψηφοφορία. Λοιπόν, 26 Ιανουαρίου η ψηφοφορία Λοιπόν, τέλος εδώ της συνεδρίασης της Επιτροπής. Από εδώ και πέρα συντονιστές. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Παρακαλώ όμως τους συντονιστές να μην φύγουν και να μην καθυστερήσουμε. Εμείς σαν Επιτροπή θα τα πούμε αύριο στις 9.